Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, άρχισε η συνεδρίαση. Χτες ο πρόεδρος ανακοίνωσε μια ερμηνεία του άρθρου 166, 167 παράγραφος 1 και 195 εδάφου 3 του εσωτερικού κανονισμού. Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συνταγματικές υποθέσεις. Εφόσον δεν έχουμε λάβει κάποια ε, αντίρρηση βάσει του άρθρου 211 του εσωτερικού κανονισμού, Θεωρούμε ότι εγκρίνεται η ερμηνεία αυτή. Μία ακόμη ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας με ενημέρωση